Μόλι δεν micro, le micro, le micro.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 Καλησπέρα σας. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ε, τρίτης ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του Πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Εγκρίθηκε. Στη συνέχεια. Πρωτοβουλία σχετικά με την Τραπεζική Ένωση. Εγκρίθηκε. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 εγκρίθηκε. Η ανατολική εταιρική σχέση εγκρίθηκε. Η πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια εγκρίθηκε. Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά εγκρίθηκε. Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Παράταση ορισμένων προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19. Εγκρίθηκε. ΦΕΝΤΕΡ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ιωρικής Ανάπτυξης, εγκρίθηκε. Ε, περιφερειακή, συγγνώμη. Ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εγκρίθηκε. Η παραπομπή ε, στην Επιτροπή για συζήτηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών εγκρίθηκε. Πρωτοβουλία για τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά το θάνατο του George Floyd εγκρίθηκε. Η πρωτοβουλία για το νόμο περί εθνικής ασφάλειας ε, της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας για το Χονγκ Κόνγκ και ανάγκη να υπερασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κόνγκ εγκρίθηκε. Η κατάσταση στο χώρο Σέγγεν μετά την εξάπλωση της επιδημίας COVID-19 εγκρίθηκε. Και τέλος, η ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 εγκρίθηκε. Έτσι έχουν λοιπόν τα αποτελέσματα του τρίτου και τελευταίου γύρου ψηφοφορίας για σήμερα. Στις οθόνες βλέπετε τις λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων ε, για τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν. Τα πρακτικά ε, της Συνόδου θα υποβληθούν στην επόμενη Σύνοδο της Ολομέλειας και αν δεν έχετε αντίρρηση θα διαβιβάσουμε τα κείμενα αρμοδίως. Τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβεστούν στα πρόσωπα και τους οργανισμούς που αναφέρονται ως αποδέκτες. Ε, βλέπω ότι δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο, οπότε ε, διακόπτεται ε, η συνεδρίαση και η περίοδος συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλό σας βράδυ.